ότι έχουν εγκριθεί. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι για την δυνατότητα που έχω να χαιρετήσω την παρουσία υψηλού επίπεδου αντιπροσωπείας του Τουνησιακού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στα θεωρία. Καλώς ήλθατε κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει, επαναλαμβάνει στα γαλλικά ο πρόεδρος της ε, συντακτικής συνέλευση της ε, Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είστε μια μεγάλη ελπίδα για όλου μα. Ich begrüße eine Delegation der Europaschule aus Ückle auf der Besuchertribüne. Es sind Schülerinnen und Schüler, die sich mit großem Einsatz für ein Schulprojekt in Sambia engagiert haben.